Μακροοικονομική βοήθεια προς το χασιμετικό βασίλειο της Ιορδανίας. Η κυρία Νέιτς έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι συγγήτρια για το σχέδιο έκθεσης Επιτροπής μας ε, προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Θα πω δύο λόγια. Έχουμε 20 τροπολογίες επί της, του σχεδίου του κειμένου μου στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη δουλειά τους. Συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες εκτός από την 14, την κυρία Λογόν Τάσεν, από τις κάτω χώρες, από το PVV της κάτω χώρες. Δεν υποστηρίζω την τροπολογία της γιατί είναι εντελώς αρνητικές και ουσιαστικά πετάει όλη την ιδέα του να δώσουμε βοήθεια στην ε, Ιορδανία. Είναι εναντίον. Φαντάζομαι ότι θέλει να την τιμωρήσει επειδή είναι μουσουλμανική χώρα. Θέλω οι συνάδελφοι τη ΣΥΝΤΑ και, του προϋπολογι... και της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού να συζητήσουν, ε, δεν θέλω μάλλον να συζητήσουν παλιότερες πτυχές του προϋπολογισμού που είναι σημαντικές, αλλά εδώ εμείς ως Επιτροπή ε, Εξωτερικών θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ορτανή να πάρει αυτή την οικονομική βοήθεια σε αυτή την ε, χαλεπή περίοδο για δύο λόγους. Καταρχάς, υπό την Αγία του Βασιλιά της Ιορδανία ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν βρίσκουν όλους σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, γιατί υπάρχουν κομμάτι του πληθυσμού που θα ήθελα να παραμείνει το status quo. Πιστεύω λοιπόν ότι για να προωθηθούν αυτές οι εξελίξεις καλό είναι να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε αυτή τη μεταβατική κατάσταση και η μετάβαση αυτή είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γίνεται με ειρηνικό τρόπο. Επίσης, δεύτερον, η Ιορδανία αντιμετωπίζει μεγάλη ροή προσφύγων από τη Συρία λόγω της σύγκρουσης στη Συρία. Και αυτός ο κόσμος, αυτοί οι μετανάστες, αυτοί οι πρόσφυγες πιέζουν δημογραφικά τη χώρα, πιέζουν οικονομικά τη χώρα και φαντάζεστε ότι και οι ίδιοι οι Ορδανοί δεν είναι πάντα ευχαριστημένοι με τις τεράστιες αυτές ροές προσφύγων αρχές της Ιορδανίας κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες βέβαια αυτούς, αλλά η κατάστασή τους είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζονται οικονομική υποστήριξη και πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο και συνετό η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει αυτή την πρόταση και το σχέδιο συμφωνίας. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς για τη δουλειά που κάνατε από αυτής της και τώρα θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές να παρέμβουν. Δεν βλέπω κανένα. Υπάρχει και ο εκπρόσωπος Κομισιόν παρόν. Ο κύριος Τεμπράνο Αρόγιο. Θέλει να πει δυο λόγια ίσως. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της και την υποστήριξη της πρότασής μας. Ε, συμφωνούμε απόλυτα με τα επιχειρηματά της. Η κατάσταση στην Ιορδανία ε, επιδεινώνεται γιατί η βασική λόγη η Συριακή κρίση καθώς και η ε, αστάθεια στην Χερσόνησο του Σινά επιδεινώνονται λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο. Και η, Αίγυπ... η, Συρι... Συγγνώμη, Ορδανία αναγκάστηκε το πετρέλαιο αυτό το οποίο δεν παίρνει πια από την Αίγυπτο ε, και που σταμάτησαν οι εισαγωγέ από τον Ιούλιο ε, να το αντικαταστήσει με το ακριβότερο φυσικό αέριο. Και αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου ε, των τρεχουσών πληρωμών αυξήθηκε στο 18,5% και υπάρχει και επιβάρυνση του ΑΕΠ κατά 10%. Επομένω, θέλουμε να δώσουμε αυτή τη χρηματοοικονομική βοήθεια. Είναι σημαντικό επίση για την αξιοπιστία τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη διαδικασία μετάβασης της Ιορδανίας. Τώρα, για τις ε, συγκεκριμένες τροπολογίες θα εστιάσω σε μία που είναι η πέντε που μιλάει για τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την Ιορδανία και που αναφέρει από ό,τι φαίνεται ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη συνεργασία ε, και την ε, δημοκρατική, το δημοκρατικό εξυγχρονισμό κτλ, πολιτική σταθερότητα ε, προφανώς θα πρέπει να το... Και, και λέω ότι μάλιστα ότι αυτό είναι ε, κριτήριο επιλεξιμότητα. Φυσικά είναι καλή η μετάβαση προ τη δημοκρατία, αλλά έτσι όπω το είναι διατυπωμένο ω κριτήριο επιλεξιμότητα, είναι αρνητικό. Επιπλέον, η χώρα αυτή, η Ορδανία, είναι χώρα που καλύπτει την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Να αλλάξετε λοιπόν την ε, διατύπωση. Στην τροπολογία 4 λέμε ότι υπό την αιγίδα τη αυτού μεγαλειότητα του βασιλιά. Έχει νόημα να αναφερθούμε σε ένα άτομο ή σε ένα θεσμό. Δεν έχουμε βασικό πρόβλημα, αλλά η διατύπωση. Επίσης, είναι σημαντικό να προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να χορηγήσει πραγματικά αυτή την οικονομική βοήθεια στην Ιορδανία. Αυτή η βοήθεια ε, ζητείται και δικαιολογείται εν μέρη λόγω της έλευσης ε, πολλών προσφύγων λόγω της Συριακής κρίσης. Επίσης θα πρέπει να θεωρηθεί, θεωρηθεί ως τμήμα της συνολικής παρουσίας και απόκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Τεμπράνο Αρόγιο. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο γνωμοδότης θα ψηφιστεί στην ε, Επιτροπή μας στις 10 Οκτωβρίου. Ήταν το τελευταίο σημείο για το πρωί. Καλή όρεξη. Θα τα πούμε το απόγευμα.